Okay, friends. Αγαπητοί φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης, έγκριση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγκρίνεται δηλαδή το σχέδιο ημερησίας διάταξης τα πρακτικά της συνεδρίασης της 3ης Σεπτεμβρίου 2014. Uh, uh, Ανακοινώ σημείο 2. Είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες πλην των Φιλανδικών, των Κροατικών και των Μαλτέζικων. Τα κροτικά επίσης, όπως ξέρετε, δεν εντάσσονται στο γλωσσικό καθεστώς επιτροπής μας. Υπάρχει μια αλλαγή στους αναπληρωτές. Ο κύριος Κάρλος Χιμένες παρετήθηκε και η κυρία Τάνια Γκονζάλη Πένας ορίστηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναπληρώτρια στην Επιτροπή απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι ο Τόμας Εντόσκι πάβει να ένα πραγματικό μέλος στην Επιτροπή μας. Τρίτον, έχετε την ε, εφαρμογή για την ψηφιακή υπογραφή στη διάθεσή σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να υπογράφετε τις τροπολογίες ηλεκτρονικά. με μια smart card ή ένα pin. It has to do with security, mobility. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής υπογραφής, ασφάλεια, κινητικότητα. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως την ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να κάνετε ατομικά αίτηση για να πάρετε PIN ή αυτή τη λεγόμενη smart card. Και όλες οι σχετικές πληροφορίες αλλά και ο σύνδεσμος για το που μπορείτε να ζητήσετε τον κωδικό PIN, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στην σελίδα μας για την Επιτροπή Απασχόληση στο e-committee. Και εκεί θα βρείτε και οδηγίες για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ε, υπογραφή, αλλά θα υπάρξει και μία ενημέρωση το Νοέμβριο. Θα σας σταλεί σχετική πρόσκληση με email. Αν έχετε ρωτήσεις, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Αντιρρήσει δεν βλέπω να υπάρχουν, αλλά μπορούν να εγκριθούν τα πρακτικά χωρί τροποποιήσει. Οπότε φτάνουμε στο σημείο 4 τη μερσιά διάταξη πτυχέ τη απασχόληση και κοινωνικέ πτυχέ τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Το 2010 ο αριθμός των πολιτών που είναι άνεργοι ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμη 16 εκατομμύρια πολίτες είναι απαραίτητο να ε, βρουν θέση εργασίας ώστε να φτάσουμε το στόχο της στρατηγικής του 2020 για 75% απασχόληση. Άρα 16 εκατομμύρια πολίτες επιπλέον. Επίσης υπάρχουν αποκλίσεις ε, στα ποσοστά απασχόλησης και αυτά μάλιστα αυξάνονται, τα, αυξάνονται αυτές οι διαφορές και μεταξύ κρατών και μεταξύ περιφερειών. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε και κινδυνεύει να δημιουργήσει αυξημένες κοινωνικές ανισορροπίες μακροπρόθεσμα αυτό το φαινόμενο. Εξού και εκ μέρους της Επιτροπής μας ε, έχω καταρτήσει μια σειρά από προφορικές ερωτήσεις προς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για να μας απαντήσουν πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Όλες αυτές τις προφορικές ερωτήσεις τις έχετε στο φακελό σας. Μπορώ αν θέλετε να σας αναφέρω ορισμένες από αυτές. Αν συμφωνήσει, μου λέγει και η Κομισιόν ότι η οικονομική κρίση από κοινού με την δημοσιονομική εξυγία σχέση αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων απασχόληση και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής 2020 είναι το πρώτο ερώτημα. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι γιατί δεν ε, μπορεί στις συστάσεις αναχώρα η Κομισιόν να ζητά από τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν, να έχουν πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις στα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα εφόσον οι περισσότεροι στόχοι αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν ε, για την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής ε, του 2020 και τρίτον, τρίτη ερώτηση, αν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει η Κομισιόν τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την επίτευξη ακριβώς των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων της ε, στρατηγικής 2020. Τέταρτον, αν Συμβούλιο και Κομισιόν ή Κομισιόν τέλος πάντων συμφωνούν ότι η απασχόληση και η μείωση της στόχιας είναι στόχοι που θα πρέπει να καταστούν ως το δυνα... μάλλον εξίσου δεσμευτικοί με αυτούς της δημοσιονομικής εξυγίανσης ώστε οι κοινωνικέ παράμετροι να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις μακροοικονομικές. Και ένα τελευταίο πώς σκέφτεται το Συμβούλιο να αυξήσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχηλοποίηση υλοποίηση στρατηγικής Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης 2020. Επίσης, έχω καταρτήσει και ένα σχέδιο ψηφίσματος, στο οποίο ακριβώς αυτά τα ζητήματα θίγω. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις θα δώσω μέσω στο λόγο ε, σε όποιον θέλει. Ο κύριος Σίμων είναι ο πρώτος. Okay. Sorry. Ε, I'll start with the Όχι, λάθος. Πρέπει να ξεκινήσω από τους συντονιστές. Ευχαριστώ. Από τη σκοπιά των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών για μας το σχέδιο είναι καλό και τρία ζητήματα παίζουν εδώ ρόλο για μας. Πρώτο, το βαθμολόγιο για τα κοινωνικά και την απασχόληση. Αυτό οφείλει να γίνει διακόπτη. Δεν υπάρχει μετάφραση προς τα αγγλικά, διαπιστώνει ο κύριος Ευρωβουλευτής. Υπάρχει πρόβλημα με τα αγγλικά, κάνει νεύμα καταφατικό. Ας αρχίσουμε ξανά λέω λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες θεωρούμε ότι το πρώτο αυτό σχέδιο είναι πολύ θετικό. Τρία ζητήματα μας απασχολούν πολύ. Πρώτο, το βαθμολόγιο, το scoreboard δηλαδή για τα κοινωνικά και την απασχόληση θα πρέπει να γίνει δεσμευτικό. Η ΔΕΜΗ δεν πρόκειται να δούμε κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη. Δεύτερο, πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι κοινωνικές επενδύσεις να αποκλειστούν από τα όρια του ελλείμματος. Μας τα έχουν δηλώσει αυτά και εξωτερικοί οργανισμοί. Η πολιτική λιτότητας δεν μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Τρίτο, χρειάζεται πολιτική απασχόληση, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής στις χώρες μέλη. Η στόχοι για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι το ίδιο σημαντική όπως η στόχη για τη δημιουργία απασχόλησης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ντάβιντ, εσείς. Όχι, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θα καταθέσουμε εν ευθέτω χρόνο τις τροπολογίες μας. Μόνο αυτό ήθελα να πω. Κύριε Κάζα, σας ευχαριστώ. Μακιντάιρ. Άλλος κανείς για τους ECR. Εσείς κυρία μου, αλλά δεν μπορώ να πω καλά το όνομά σας. Κυρία Χάρκιν, Χάρκιν, αυτό είναι το σωστό όνομα, ορίστε. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, γιατί και εμείς θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες, ερωτήσεις. Παράγραφος 7. Λέμε και αμοιβαία συμφωνημένες συμβατικές ρυθμίσεις. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει αμοιβαία αποφασισμένες ή εγκεκριμένε συμβατικές ρυθμίσεις. Δεν καταλαβαίνω καλά. Επίσης, παράγραφο 9. Αύξηση επενδύσεων στις υποδομές. Εκεί να μπει βέβαια και έρευνα και ανάπτυξη, πράσινες θέσεις απασχόλησης κλπ. Δέκα. Λέμε για αποκλεισμό ορισμένων επενδύσεων από τους εθνικούς λογαριασμούς. Θα είναι δύσκολο να συμφωνηθεί αυτό, να υπάρχει συμφωνία δηλαδή σε αυτό. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες. Για την παράγραφο 15 τώρα. Εκεί μιλείται για ένα δίκτυο που θα αφορά την σχετική φτώχεια. Εδώ χρειάζομαι κάπως περισσότερες εξηγήσεις. Εγώ βέβαια καταλαβαίνω τι σημαίνει, αλλά δεν είμαι βεβαία ότι υπάρχει τέτοιος δείκτης και αν έχει χρησιμοποιηθεί κάποτε στο παρελθόν. Εκτός από αυτά, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι για τις προφορικές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια για τις πτυχές απασχόλησης και κοινωνικές για την Ευρώπη του 2020 στις ερωτήσεις 1 και 4. Αντί να πούμε συμφωνεί η Επιτροπή, να πούμε καλύτερα θεωρεί η Επιτροπή. είναι ένας διαφορετικός τρόπος διατύπωσης, αλλά έχει σημασία. Αυτά είναι τα σχόλια που είχα να κάνω. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ. Για λογαριασμό της δικής μου πολιτικής ομάδας, της Ενωτικής Αριστεράς, θέλω να υποστηρίξω και εγώ το σχέδιο. Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες που βάζει είναι σωστές και καθιστά σαφές επίσης ότι η απασχόληση και ιδίως η ποιοτική απασχόληση και η καταπολέμηση της φτώχειας πάνε χέρι με χέρι. Γι' αυτό άλλωστε συμφωνώ την κατανομή των, στην κατανομή των θεμάτων και υπενθυμίζω στην κυρία Χάρκιν διότι ρωτήσατε πριν στην παράγραφο 15, παράγραφο 15 για τον δίκτυ της σχετικής φτώχειας. Στην προηγούμενη Ευρωβουλή είχαμε κάνει τη συζήτηση αυτή κατ' επανάληψη και σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνία και έχει τοποθετηθεί για την σχετική φτώχεια, έχει εξηγήσει τι εννοεί, πρόκειται για τον δίκτυ που λαμβάνει υπόψη τους μέσους μισθούς και τα μέσα εισοδήματα των οικοκυριών εθνικά και υπενθυμίζω ότι και στα πλαίσια του, έτους, ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας, τα είχαμε πει αυτά. Εκεί αναφέρεται η παράγραφος 15, ότι στο μέλλον δηλαδή οι χώρες μέλη μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς δείκτες. Αυτό που ζητείτε εδώ είναι να επανέλθουμε σε μια κοινή βάση δεδομένων, σε μια κοινή λήψη υπόψη δηλαδή, της βάσης δεδομένων και ο δείκτης να μπορεί να λαμβάνει υπόψη ανά πάσα στιγμή. Είναι σημαντικό όμως οι χώρες μέλη να διακρίνουν ανάμεσα σε μήλα και αχλάδια, τι θέλουν να κάνουν τέλος πάντων και με ποιο τρόπο θα επιδιώξουν να επιτύχουν τους στόχους. Ε, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Jim Lambert. thank you. Thank you, President. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο-τρία από τα δικά μου σχόλια τα ε, είπε μόλις πριν η κυρία Χάρκιν. Αλλά στις ερωτήσεις, τις προφορικές, νομίζω θα πρέπει να πούμε κάποια λόγια για τις επενδύσεις και συγκεκριμένα ότι θέλουμε να επενδύσουμε σε τομείς που θα μπορούσαν ε, δυνητικά να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στο μέλλον και στόχος μας είναι να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και ευχαριστώ για την ενεργειακή απόδοση, για το φωτισμό. Λοιπόν, στο ψήφισμά μας τώρα, επειδή θα μας απασχολήσουν πιο πολύ κοινωνικές πτυχές και η πτυχή της απασχόλησης ως Επιτροπή. Ε, καταλαβαίνω την εστίαση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και μια διασύνδεση με τις άλλες διαστάσεις της ε, σταδικής 2020, όχι μόνο την ε, ανάπτυξη για όλους, αλλά και τις άλλες δύο πτυχές, βιώσιμη και ευφυής και νομίζω ότι θα πρέπει οι τροπολογίες μας ε, προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα την παράγραφο 15 για τους δείκτες για τη φτώχεια, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά από το δίκτυο ελάχιστου εισοδήματο, το οποίο δίνει συμβουλές όχι μόνο για ένα ε, δείκτη, αλλά για δύο, δηλαδή και τη σχετική και την απόλυτη φτώχεια, γιατί σε κάποια κράτη-μέλη η απόλυτη φτώχεια είναι ένα δείκτης που ακόμη ισχύει. Σίγουρα έχουμε επισημάνει, το είπε και η Γκάμπι Τσίμερ, ότι έχουμε απορίες σε σχέση με τις επιλογές των κρατών μελών για τους δείκτες. Άρα θα καταθέσουμε σίγουρα τροπολογίες ε, επ' αυτού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κ. Σάιμον. Ευχαριστώ. Πολλές φορές ε, υπάρχουν ε, πράγματα μεγάλα που είναι τόσο λάθος, αλλά είναι τόσο μεγάλα που δεν έχει νόημα ίσως να συζητούμε για αυτά πια. Ε, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να τα συζητούμε συνεχώς και πρέπει να σας πω ότι το κριτήριο του χρέους και το κριτήριο του ελλείμματος είναι νομικά δεσμευτικά ε, και συνδέονται με κυρώσεις. Πολύ εχμηρές, πολύ ε, σημαντικές. Ενώ οι διαστάσεις για τη στρατηγική 2020 έχουμε απλά εκεί στόχους, ε, φιλοδοξίες. Είναι μια στρατηγική. Ούτε κυρώσεις έχουμε. Και αυτό είναι άδικο, θεμελιωδώς. Η Ένωση αυτή δεν χαρακτηρίζεται από ισορροπία, έχει πουλήσει κατά κάποιο τρόπο τους πολίτες της, γι' αυτό και δεν την εμπιστεύονται πλέον. Βλέπουμε δηλαδή ότι πόσο τα ψηρίζουμε όλα για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, αλλά όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές πρακτικές, δεν ισχύει το ίδιο. Thank you, Mr. Simon. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σάιμον. Πυρίνσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γιατί την παράγραφο 10 του σχέδιου ψηφίσματος θέλω να κάνω ένα σχόλιο, το είπε και η κυρία Χάρκιν όταν ε, έκανε τα σύντομα σχόλιά τη, υπό την έννοια ότι η ιδέα τη εξαίρεση ορισμένων επενδύσεων από τον υπολογισμό των εθνικών ελλημάτων είναι πολύ δύσκολο ή μάλιστα θα έλεγα και αδύνατο ε, να τύχει συμφωνίας. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να είμαστε στο δυνατόν πιο ευέλικτοι στις προτάσεις μας. Συγκεκριμένα έχω καταθέσει και μια τροπολογία για την παράγραφο 13 που λέει ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, επενδύσεις επίσης σε επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι από το από τους στόχους αυτό το οποίο εξαιρείται είναι η καθαρή αύξηση των δημόσιων δαπανών στους ανωτέρω ε, τομείς πολιτικής στόχους. Και αυτό να γίνεται σε τέτοια βάση. Νομίζω ότι έτσι αντιμετωπίζεται και ε, η ανησυχία ότι αφήνουμε πόρτα ανοιχτή σε μία είδους ανευθυνότητα ε, για την κατάρτιση του προπολογισμού και κάποιες αυθαίρετες, κάποιους αυθαίρετους αποκλεισμούς ή εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάποιες στόχοι που ήδη έχουμε συμπεριλάβει με βάση το, το έτος αναφοράς καλό τους συναδέλφους να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς, ε, ναι, μεν μιλάμε για πολιτικές και για επενδύσεις, αλλά εάν δεν είμαστε ευέλικτοι και στο τεφα του στόχου του δημοσιονομικού ελλείμματος, θα μείνουμε στα λόγια. Ευχαριστώ. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστώ. Κύριε Σμάν. Α, μόλις εκαλύφθην. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Η κυρία Σάντερ. Στο σχέδιο ψηφίσματος ε, αναφέρονται διάφοροι δρόμοι για να μειωθεί η φτώχεια των νέων και ο αποκλεισμό. Εγώ πιστεύω πως ίσως λείπει μια παράγραφος που θα θυμίσει ότι ευνοώντας ένα νομικό πλαίσιο, κυρίως ε, την επιχειρηματικότητα ευνοώντας, ε, θα μπορούσε και αυτό να είναι ένας δρόμος για αυτούς. Να ευνοήσει δηλαδή την κατάσταση των νέων. Ευχαριστώ, you. Ε, Mr. Ε, Ο κύριος ε, Μάλιστα, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την παράγραφο 7. Είναι αλήθεια πως κάτι δεν κατάλαβα εκεί. Πρόκειται για μία ε, συμβατική κατάσταση ανάμεσα στις κυβερνήσεις και την Κομισιόν ώστε να αναλάβουν την υποχρέωση διαρθωτικών αλλαγών, πράγμα που θα τοποθετούσε το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια στην άκρη. Εν πάση περιπτώσει, αν διαβάσει κανείς αυτή την παράγραφο, μπορεί να καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Δεν αναιρεί τη στήριξη αυτού του κειμένου, αλλά πάντως υπάρχει μια φυσιμία που θα πρέπει να εμβαθύνουμε για να καταλάβουμε ακριβώς περί τι πρόκειται. Δεύτερη παρατήρηση και θα σταματήσω. Θέλω να αναφερθώ σε μια παρέμβαση που έγινε και φορούσε τις επενδύσεις, ότι δηλαδή αυτές στο μέλλον θα πρέπει να καταγράφονται ε, και να διέπονται από ε, δεσμευτικά κριτήρια. Θα πρέπει να δούμε τι λέγεται από την διεθνή δηλαδή οι διεθνείς ε, οργανισμοί που δεν χαρακτηρίζονται αριστεροί, αριστεροί όπως ας πούμε το Δούνο του, που δεν πάβει να λέει πως αν σήμερα μπορούν εκείνοι να στηρίξουν κάποιες διαστατικές μεταρρυθμίσεις, εάν δεν αντισταθμιστούν από ε, μαζικές επενδύσεις, είναι, θα, θα μπούμε σε ύφεση. Ο Μάριο Ντράγκη δεν λέει τίποτα άλλο γιατί το να εκδίδει χρήμα είναι πολύ ωραία για μια κεντρική τράπεζα. Το θέμα είναι ποιο θα τα απορροφήσει αυτά τα χρήματα. Πάντοτε έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Έχουμε κανόνε που είναι πεπαλαιωμένοι, δεν αντιστοιχούν στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα και εμεί εδώ θα επιμένουμε στη θέση μα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ την κυρία Ούλσκοπ για το καλό αυτό σχέδιο ψηφίσματος. Η Ευρώπη 2020 είναι η στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην αποτύχει αυτή η Ευρώπη 2020, όπως απέτυχε η Λισαβόνα. Ανάπτυξη λοιπόν. Εμείς έχουμε πάντα βάλει πέντε βασικούς στόχους. Απασχόληση, έρευνα, ανάπτυξη, κλίμα ενέργεια, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας. Έχουμε και 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες για την ψηφιακή οικονομία, την νεότητα, τη βιομηχανική πολιτική, την καταπολέμηση της φτώχειας και την αποδοτική χρήση των πόρων ενέργειας. Η προσπάθεια για την Ευρώπη 2020 θα ξεκινήσει από την ενιαία αγορά. Με πιο πολλή δουλειά. Αυτά πρέπει να απηχούνται και στις κοινωνικές πτυχές της, απασχόλησης, της ε, ε, πολιτικής αυτής, που πρέπει να είναι συμπληρωματική η στόχη αυτή, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε την κοινωνική εκείνη προστιθέμενη αξία που επιθυμούμε. Ως Ευρωπαίος Βουλευτής, τονίζω ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία του δημογραφικού παράγοντα που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Πληθυσμός που γυράσκει, μείωση των γεννήσεων, διαφορετικές δομές της οικογένειας. Ήδη από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έγγραφο στρατηγική έχει υποσχεθεί να λάβει υπόψη και να εξασφαλίσει καλύτερους όρους υπέρ των οικογενειών και την καλύτερη διασύνδεση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Τα θεωρεί αυτά δε ως είπα τους στόχους. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσανατολιζόμαστε εκεί. Ο συντονισμός της οικογενειακής πολιτικής μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής οικογενειακής στρατηγικής, στρατηγικής για την οικογένεια δηλαδή για να εξασφαλιστεί έτσι η επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Θα χαρώ πολύ αν επιτύχουμε όλοι μαζί να λάβουμε περισσότερο υπόψη τον παράγοντα της δημογραφίας και να τον τονίσουμε περισσότερο στο σχέδιο ψηφίσματος. Thank you. Is there anyone from Ευχαριστώ. Από την Κομισιόν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. No. Uh, well, um, uh, Σας ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο προφορικής ερώτησης. Και όσον αφορά την παράγραφο 7, νομίζω ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε και θα το πράξουμε όντως. το ψήφισμα και η προφορική ερώτηση θα, οι προφορικές ερωτήσεις θα υποβληθούν σε αυτό το χρόνο εξ ονόματος της Επιτροπής μας για την Ολομέλεια της, ε, του Νοεμβρίου. Και λόγω χρονικών περιορισμών οι τροπολογίες θα μπορέσουν να κατατεθούν μόνο από τους συντονιστές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και αν γίνεται στα αγγλικά μόνο. just give you Να σας δώσω λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Τα έγγραφα υπάρχουν υπάρχουν διαθέσιμα στο 84 AM. Ίσως είναι πιο εύκολο για σας. Η προθεσμία για τους συντονιστές είναι η 7η Οκτωβρίου. Η εξέταση αυτών των τροπολογιών στα αγγλικά, όπως είπα, το υπογραμμίζω ξανά, είναι η 16η Οκτωβρίου. Τώρα, η έγκριση στην Επιτροπή από, ε, Απασχόλησης εδώ θα είναι στις 4 και μετά θα έρθει στην Ολομέλεια στις 24 με 27 Νοεμβρίου. Αυτό είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Και μάλιστα όπως υπογραμμίσατε πρόκειται για πολύ σημαντική πολιτική δήλωση από την Επιτροπή Απασχόλησης. και σας ευχαριστώ θερμά για τις παρεμβάσεις γιατί όντως ε, ε, περί αυτού πρόκειται. Είμαστε πολύ πιο μακριά από αυτό που αναμέναμε όταν ε, αποφασίσαμε για τη στρατηγική 2020. Yes, you wanted the floor. Μάλιστα, θέλατε το λόγο. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλά θα ήθελα να σας πω με βάση τα όσα ακούσαμε, πραγματικά με σοκάρει σημείο πρώτον το, ότι οι τροπολογίες δεν επιτρέπονται μόνο για τους, συντονισμένους, ε, για τους συντονιστές, άρα οι μη εγγεγραμμένοι δεν μπορούν να εκφραστούν και δεύτερον ότι επιτρέπεται μόνο τα αγγλικά. Πράγμα το οποίο είναι δεσμευτικό για όσους δεν γνωρίζουν την αγγλική και κυρίως γιατί πολύ συχνά είναι τρελέ οι, οι προθεσμίες, δηλαδή τις παίρνουμε την παραμονή για την επομένη. Ε, ε, ε θέλουμε όμως να είμαστε νόμιμοι απέναντι σε όλους μα τους συμπολίτες, σε, σε όλες τις χώρες της Ένωσης, αλλά αν δεν μπορούμε να δουλέψουμε, εδώ δεν αξίζει τον κόπο καν να ερχόμαστε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσίμερ. Συμφωνώ ότι και εγώ εξεπλάγει και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι απόφαση των συντονιστών. Θα πρέπει να το είχαμε πληροφορηθεί. Εγώ ξέρω αγγλικά, μπορώ να γράψω τις τροπολογίες ε, στα αγγλικά, αλλά δεν κατάλαβα. Ε, ε πρέπει να ενημερωνόμαστε ε, εκ των προτέρων αν μόνο οι συντονιστές πρέπει να υποβάλουν το προγείες, αν πρέπει να είναι μόνο στα αγγλικά, πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πού προήλθε αυτή η απόφαση, γιατί με εξέπληξε. Ναι, για όλους μας είναι εκπληκτικό, αλλά θέλουμε να επηρεάσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή πριν να λάβουν απόφαση. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δουλέψουμε τόσο γρήγορα. Εάν θέλουμε απλά να διατυπώσουμε κάτι που πιστεύουμε, τότε μπορούμε και να έχουμε άλλο χρονοδιάγραμμα. Εάν θέλετε όμως να επηρεάσουμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν, τότε οφείλουμε να δουλέψουμε με αυτό το ρυθμό. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να δουλέψουμε λοιπόν σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα και όσον αφορά τους μη εγγεγραμμένους, εσείς μπορείτε βεβαίως να υποβάλλετε τη δική σας συμβολή, αλλά πάλι στα αγγλικά παρακαλώ γιατί διαφορετικά δεν θα προκάνουμε. Και βέβαια τα σχόλια σας θα είναι στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Αν θέλετε να είναι κάτι παραπάνω από συζήτηση, αν θέλετε να είναι κάτι που να έχει αντίκτυπο στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν, τότε πρέπει να βιαστούμε και να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτά έχει η ζωή. Ε, item 5 ε, on the agenda. Σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 είναι ψηφοφορίες. While we are looking for our... Ενώ όλοι ψάχνουμε τις κάρτες μας, μπορείτε να πάρετε το λόγο αν θέλετε. Να δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή, τον κύριο Σέρχιο Γκουτιέρεθ Πριέτο Και μετά θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις των σκιωδών. Κύριε Πριέτο. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας παρουσιάσω αυτές τις συμβιβαστικές προτάσεις. Πράγματι, Είχαμε μια πρώτη έκθεση θα έλεγα, δύο από τις σημαντικότερες εκθέσεις που εκπονεί η Επιτροπή μας για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το Φεβρουάριο και τώρα για τις ε, συστάσεις αναχώρα. Και στην πρώτη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή είπαμε ότι είναι ανάγκη να εκπέμψουμε ένα ηχηρό μήνυμα από την Επιτροπή μας προς τις άλλες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βέβαια κυρίως προς τα άλλα θεσμικά όργανα σε σχέση με τις ε, κατ' εμάς προτεραιότητες ή βασικές ε, ε, κατευθύνσεις του έργου μας για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων με ευγνώμων για την συνεργασία που είχαμε. 36 είναι οι συμβιβαστικές προτάσεις που καταθέσαμε και αυτό δείχνουν πόσο πολύ προσπαθήσαμε να έχουμε διάλογο, διαπραγματεύσει, συνένεση. Και όπως είπα, θελήσαμε να θεσπίσουμε τις γενικές κατευθύνσεις για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρώτα απ' όλα, ε, εκδηλώνουμε την ανησυχία μας για το ότι ναι, δεν υπάρχει μια εύθραυστη κοινωνική ε, ανάκαμψη. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες. Έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, άνευ προηγουμένου. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πρόβλημα ποιότητας επίσης εργασίας. Πολλές φορές δηλαδή δεν μπορούν

Ε, να φύγουν από την λεγόμενη εργασιακή φτώχεια, όπω την αποκαλούν ορισμένοι οικονομολόγοι ή συμπολίτε μα και σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερε προσπάθειες για τόνωση τη απασχόλησης και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασία. Επίση, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε ώστε οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει που ζητούνται να είναι μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη ανταγωνιστικότητα ε, στην οικονομία μα, ε, τα κοινωνικά πρότυπα να παραμείνουν παραμείνουν υψηλά, κάτι που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και βέβαια να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στην καινοτομία που είναι η καλύτερη εγγύηση για να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία που όμως ε, θα διατηρεί όπως είπα και τα κοινωνικά της πρότυπα. Ζητούμε επίσης οι εργασιακέ μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν να ε, διορθώσουν μεταξύ άλλων και τις ε, μεγάλες ε, ανισότητες και τον κατακαιρματισμό, τη διάσπαση που έχουμε στα συμβόλαια, στη συμβάση, ιδίως ό,τι αφορά τη γυναική απασχόληση και την απασχόληση των νέων. Ζητούμε επίσης να συμμετάσχουν όλοι οι επιτροποί, το Σώμα των Επιτρόπων, ε, στην κατάρτιση μιας εγκάρσιας ε, πολιτικής και μιας φιλόδοξης στρατηγικής που ζητούμε από την Επιτροπή Απασχόλησης εμείς εδώ, για να έχουμε αξιοπρεπή εργασία για απασχόληση για τα επόμενα χρόνια και θεωρούμε ότι γι' αυτό δεν θα πρέπει την πολιτική να την κατευθύνει μόνο ο Επίτροπος Αρμόδος για την Απασχόληση, αλλά να είναι μια πολύ φιλόδοξη πολιτική και να ε, την συνδιαμορφώνουν ε, όλοι οι επίτροποι. Επίσης αναφέρουμε συγκεκριμένα προβλήματα που μας ανησυχούν και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες από τα κράτη-μέλη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, ε, την νεανική ανεργία, ανεργία των νέων αλλά και τους μακροχρόνια ανέργους. Ε, που πραγματικά δημιουργεί ένα ανησυχητικό θύλακα φτώχεια ε, που δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ του συναδέλφου γιατί όλε οι πολιτικέ ομάδε βοηθήσαμε να υπάρξει ε, συμβιβασμό ό,τι αφορά την κοινωνική ένωση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων να μην χάσει την προοπτική και τον ορίζοντα. αυτό ο κοινωνικός πυλώνας, το κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο δεν πρέπει να χαθεί παρά τις δυσκολίες, παρά τις δύσκολε οικονομικέ συγκυρίε που βρισκόμαστε. Και κυρίως θέλω να πω ότι είμαι περήφανος για τις ε, συμβιβαστικέ που έχουμε για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την ε, πολιτική επανεκβιομηχάνησης που απαιτείται αν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια ότι έχει να κάνει με τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Είναι κάτι που το διεκδικούμε για την οικονομική διακυβέρνηση, τον συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών. Πρέπει δηλαδή οι πολίτε να θεωρούν ότι ταυτίζονται γιατί του εκπροσωπεί και το, Εθνικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια σε αυτή την όλη διαδικασία. Έχουμε τον κανόνα 54 ε, για την Οικονομική Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι συνενετική έκθεση από προϊόν διαλόγου, προϊόν διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι μπορεί να εκφράσει ε, την άποψη της πλειοψηφία των μελών μας. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές για τη δουλειά τους και επαναλαμβάνω ήταν πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Madame Ευχαριστώ κύριε Φοντανιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα προσθέσω πολλά στα όσα μόλις είπε ο συνάδελφος Γκουτιέρεφ. Νομίζω ότι συνόψισε ουσιαστικά όλες τις τροπολογίες ε, ή τέλος πάντων τις συμμεπαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε. Θα ήθελα πολύ απλά μόνο να πω ότι τελικά φτάσαμε πράγματι σε μια μεγάλη συνένεση η ομάδα του ΕΛΚ σχεδόν, όχι όλε, σχεδόν όλε οι συμβαστικέ προτάσεις θα τις υπερψηφίσει, αλλά νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες κατέβαλαν προσπάθεια, γιατί το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε, ε, να έχουμε αυτή την έκθεση. Και φυσικά δεν είναι δική μας έκθεση, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία ε, του συμβιβασμού, να καταλήξουμε δηλαδή σε μια συμφωνία για να μπορούν να συμφωνήσουν σχεδόν όλε οι πολιτικέ ομάδε. Κάτι που πετύχαμε, πιστεύω. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τον Σέρχιο Γκουτιέρεθ. Έκανε πολλέ προσπάθειε για να πετύχει τη συνένεση. Ξέρω ότι κάποιε φορέ ίσω θα ήταν καλό να ήταν διαφορετική, σε κάποια σημεία τουλάχιστον έκθεση, αλλά και ε, με τις δικές μας υποχωρήσεις και από άλλες πολιτικές ομάδες καταλήξαμε σε μια έκθεση που νομίζω ότι μπορούμε να τη στηρίξουμε και θα τύχει της ε, ευρείας πλειοψηφίας. Ευχαριστώ. Thank you, Madam. Ευχαριστώ. κυρία Μπαντάγεβα. Oh, thank you, Chair. Um, I would also uh, thank... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια των συνεδριάσεων των σκιωδών. Η Άλτεν γέννη ευχαρίστω υποστηρίζει τι περισσότερε συμβιβαστικέ. Βέβαια, υπάρχουν κάποιε συμβιβαστικέ όπου δεν φτάσαμε ε, σε συμφωνία λόγω διαφορετικών ιδεολογικών απόψεων. Ευχαριστώ ωστόσο και πάλι για τη συνεργασία και για τα σπουδαία μαθήματα Ισπανικών που είχαμε στη διάρκεια των συνεδριάσεων των συντονιστών. Κυρία Λαμπέρτς, όχι. Ειρήνα Ρόνια Κάρι. Δεν είναι εδώ. Mr. Mann. Ο κύριος Μάν. Ναι. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Λέει εδώ συμβιβασμό, συμβιβασμό και στο τέλος λέει κατατεθειμένο από τον εισηγητή. Δεν λέει ποιες πολιτικές ομάδες συμμετέχουν στους συμβιβασμούς. Κάποιες πολιτικές ομάδες εξέφρασαν και επιφυλάξεις τώρα πριν από λίγο και είπαν ότι μετά δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν. συμφωνήσουν. Πρόκειται λοιπόν για θέση όλων των κομμάτων ή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Δεν περιλαμβάνεται αυτό στα έγγραφα. Εγώ για παράδειγμα έχω σημαντικά προβλήματα με, τις, ε, με τους συμβασμούς σίγμα και ταφ στην παράγραφο 16 που πρόκειται για τους αυτόματους σταθεροποιητές όπως η ασφάλιση των ανέργων που απορρίπτεται απολύτως σε ορισμένες χώρες μέλη. Πρόκειται για μια συζήτηση που οφείλει να διεξαχθεί. Γι' αυτό και ρωτώ πίσω από τις συμβαστικές προτάσεις ποιες ομάδες βρίσκονται. Είναι όλες, αν είναι όλες θα πρέπει αυτό να λέγεται καθαρά. Το βλέπετε στην λίστα ψηφοφορίας που έχουν ε, οι διανύμοι πολιτικές ομάδες. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στου σκιώδει εισηγητέ, που όμως δεν είναι όλοι παρόντες ή παρούσες. Όμως εσείς μπορείτε να το δείτε στη λίστα ψηφοφορία. Now we'll start the... Τώρα θα αρχίσουμε την ψηφοφορία. Αν έχετε μπροστά σας τη λίστα ψηφοφορίας, σας δίνω και λίγο χρόνο για να βρείτε τις κάρτες σας you follow, we work compromise, compromise F. Who's in favor, against, abstention, compromise. All set. Είσαστε έτοιμες και έτοιμοι. Να αρχίσουμε λοιπόν με την πρώτη, δηλαδή τη συμβαστική F. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Θέλετε... Υπάρχει πρόβλημα με το μηχάνημα. Για την ώρα ψηφίζουμε με ανάταση του χεριού. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά ηλεκτρονική επαλήθευση, οπότε θα χρησιμοποιήσετε τώρα τις κάρτες σας. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται λοιπόν με διαφορά δύο ψήφων. Τότε λοιπόν ψηφίζουμε την 37 υπέρ. Μια στιγμή υπάρχει εδώ κάποια ε, αμφισημία. Όχι, αυτή έχει εκπέσει. Η 37. Πηγαίνουμε στη 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 45 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και αυτή. 46 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ας ελέγξουμε λοιπόν με ηλεκτρονικό τρόπο ψηφίσατε τέλος τώρα της ψηφοφορίας Εγκρίνεται λοιπόν, όπως βλέπετε και στον πίνακα. Είναι καινούριο το μηχάνημα εδώ. Υπαριθμού 47 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική age ή Ήτα δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα στην παράγραφο 3 τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία καπα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 67 τώρα. Στην παράγραφο 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. μία ψήφος παραπάνω από ό,τι προβλέπεται από το Λαϊκό Κόμμα. Άρα θα πρέπει ένα αναπληρωματικό μέλος να βγάλει την κάρτα του από την σχισμή. Ωραία είναι, εντάξει, συμφωνεί τώρα. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβιβαστική λάμδα, L. Υπέρ κατά αποχές αυτή εγκρίνεται Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβιβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 78. Υπέρ, κατά, αποχές. Καλύτερα να το κάνουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψήφου. Εγκρίνεται λέει πρόεδρος, αλλά δεν φαίνεται να είναι σωστό αυτό. Όχι, απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν. Συμβιβαστική. Ευδόχη. Συμβαστική 79 πρώτα. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική νη. Εν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ο, όμικρον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενενήντα τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές ας την επαληθεύσουμε αυτήν καλύτερα τέλος και απορρίπτεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα χρειαστεί και αυτή να την παληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Τέλος της ψήφου. Εγκρίνεται λοιπόν. Λέει η πρόεδρος. Όχι, όχι, όχι. Μα είναι πράσινο το, το 24 και κόκκινο το 25. Μου φαίνεται σαν να λέει λοιπόν ότι είναι εντάξει, αλλά βεβαίω απορρίπτεται. Οι υπαριθμών 98 και 99 υπέρ κατά Ναι, νομίζω πρέπει και αυτό να το επαληθεύσουμε. πέρα της ψηφοφορίας. Τώρα είναι σωστά τα χρώματα. Το πράσινο μου τα δείχνει καλά αυτή τη φορά. Εγκρίνεται λοιπόν. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πί, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. υπαριθμών 109. 109, 10 και 11 όλες μαζί γιατί είναι ακριβώς ίδιες πρέπει να ψηφιστούν όλες μαζί ψήφι υπέρ κατά αποχές έλεγχος Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 113 υπέρ κατά Α, ναι, ναι, αυτή εκπίπτει, εκπίπτει, ωραία. Τώρα πάμε στην 114 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά Άποχες. Χρειάζεται επαλήθευση και εδώ. Πέρας. Πάλι μια υπερβάλλουσα ψήφος του Λαϊκού Κόμματος. Κάποιος να τη βγάλει. Ωραία λοιπόν. Από... 122 στην παράγραφο 14α, έτσι. 122 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική R, ρο δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή εγκρίνεται. της κυρίας Τζιν Λάμπερτ η 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική S, σίγμα, υπέρ, κατά, αποχές, Δεν είναι εύκολο λοιπόν να κάνουμε επαλήθευση ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται βέβαια, θα έπρεπε να το είχα δει και από την πρώτη φορά. Συμβαστική συμβαστική ταφ, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κύριο Σάιμον. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή Εκατόν σαράντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση, check. Ωραία, ας κάνουμε λοιπόν. Πέρας τώρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική U υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, αρχίζει η ψηφοφορία λέει η πρόεδρος, τώρα κλείνει. Περάσει τώρα τη ψυχή. Απερίφθη λοιπόν. Τροπολογία 161 υπέρ

162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας γίνει επαλήθευση εδώ. Ελεκτρονική. Τέλος. Και απερίφθη αυτή. τέσσερα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 χ δηλαδή υπέρ κατά αποχές επαλήθευση εδώ ηλεκτρονική Πέρας της ψήφου. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Συμβαστική ύψιλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι μάλλον την απορρίπτεται αλλά ας την κάνουμε και ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουρες πέρας απορρίφθηκε λοιπόν 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάντως αν θέλετε μπορούμε να την επαληθεύσουμε και ηλεκτρονικά ωραία ας το κάνουμε άρχισε η ψηφοφορία και τώρα κλείνει Εγκρίνεται σαφώς. Συμβαστική Z, Z δηλαδή, με προφορική τροπολογία. Πρώτα πρέπει να ρωτήσω αν υπάρχουν ενστάσεις κατά της προφορικής τροπολογίας που έχει καταθέσει το Λαϊκό Κόμμα. Δεν υπάρχουν ενστάσεις λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τότε την προφορική τροπολογία και ψηφίζουμε την συμβαστική ζήτα υπέρ. Κάποιος δει το λόγο. Πρώτα πρέπει να πούμε αν υπάρχει προβλήμα, κάποιο πρόβλημα γιατί με, και μετά να δούμε αν ε, δεχόμαστε να ψηφίσουμε για προφορική τροπολογία και μετά να ψηφίσουμε για τη συμβιβαστική. Μα, μα είναι ήδη στην, ε, στον κατάλογο ψηφοφορίας. Δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Την έχετε την ε, προφορική τροπολογία μέσα στην λίστα ψηφοφοριών. Μα ρωτήσατε άλλωστε εάν υπάρχουν ενστάσεις για, κατά της προφορικής τροπολογίας. Το ρωτήσατε κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κάσα. Επομένως, αφού δεν υπάρχουν ενστάσεις, τώρα ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προφορική. Βεβαίως το Προεδρείο αποφασίζει λέει ο κ. Πριέτο, εσείς αποφασίζετε, αλλά εγώ πάντα νόμιζα ότι πρώτα ψηφίζεται η προφορική τροπολογία και μετά η συμβιβαστική. Εγώ έτσι είχα καταλάβει. Ε, I'll give the floor to, to ε, ε, Jutta Steinruck. Die S&D-Fraktion ist gegen das, die mündliche, den mündlichen Änderungsantrag. Ο κύριος Κάσα. Κυρία Πρόεδρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εσείς ρωτήσατε αν υπήρχαν ενστάσεις κατά της προφορικής τροπολογίας. Τώρα προχωρείτε σε άλλη διαδικασία. Εμείς δεν συμφωνούμε, αλλά δεν μπορείτε να ανατρέψετε τη διαδικασία. Δεν μπορείτε τώρα να υποβάλλετε ένσταση για την προφορική τροπολογία. Αν θέλετε μπορείτε να καταψηφίσετε τη συμβιβαστική. If the oral is rejected, then you vote on the original text. Mm. You have two options. It's up to you. Uh, oh. Η πρόεδρος. Ας αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Υπάρχουν ενστάσεις κατά της προφορικής τροπολογίας. Χρειάζεται παραπάνω από τρεις ενστάσεις κατά της προφορικής τροπολογίας. Μπορείτε να ηγερθείτε αν θέλετε. Μπορείτε να σηκωθείτε όρθιοι. I think, Mr. Kassa, that we have... Κύριε Κάσα, νομίζω ότι βρήκαμε τη λύση. Λέει η Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε τη συμβιβαστική ζήτα με την προφορική τροπολογία και μπορείτε βεβαίως να ψηφίσετε είτε υπέρ είτε κατά, όπως επιθυμείτε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την συμβαστική τροπολογία Ζ με την προφορική τροπολογία, λέει ο κύριος Πριέτο. Όσοι λοιπόν είναι υπέρ, όσοι είναι κατά, αποχές και θα κάνουμε παρήθευση ηλεκτρονική. Πέρας, τέλος δηλαδή της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και προχωρώ. Στην 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2α, Αλφα-αλφα δηλαδή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική αβ, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC, ΑΣ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Διακόσια τέσσερα υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. πέντε υπέρ κατά αποχές Ας κάνουμε επαλήθευση. 205. Ψηφίζομαι. Τέλος. Σαφής η διαφορά. Εγκρίνεται λοιπόν. Η 206 τώρα στην παράγραφο 24 υπέρ κατά αποχές χρειάζεται επαλήθευση αυτή εδώ η ψηφοφορία. πέρασε, Εγκρίνεται πάντως. 211 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τσεκ. 211. Αρχίζει και ξανακλίνει. Α, η Γιούτα. Είχε κλείσει όμως η ψηφοφορία κανονικά, ε. Πάντως ούτως ή άλλως έχει απορριφθεί. 210 ψηφίπερ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση λοιπόν, ωραία, τσεκ, 210, αρχίζει και κλείνει πάλι. Δεν εγκρίνεται, απορρίπτεται. 207. Όχι, 212. Τροπολογία 212, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α δέλτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική e. ΑΕ, ΑΕ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί η 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AF, αφ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η AG, συμβαστική AG, στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 238. Ευχαριστώ. Ε, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική AH, αλφα ή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 242, υπέρ. 242, υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Χρειάζεται επαλήθευση εδώ. Αρχίζει. Τώρα τελειώνει. Εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 253 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται έλεγχος ηλεκτρονικός αρχίζει και τελειώνει Απορρίφθηκε. 251. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 255 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε επαλήθευση 255 αρχίζει η ψηφοφορία και τώρα λίγη και απερίφθη Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι τώρα η 7. Ακολουθεί η τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ χρειάζεται έλεγχος. Έκλεισε εδώ η ψηφοφορία, τελείωσε και απερίφθη. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ θα χρειαστεί check. Αρχίζει η ψηφοφορία και τώρα κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Καλά λοιπόν, 22. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Α, εγκρίνεται. Συμβαστική σε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία που θα γίνει ονομαστικά. Πέρας. Βλέπετε το αποτέλεσμα, 41 υπέρ, 5 κατά και συγχαρητήρια στον κύριο Κουτιέρες. The voting will proceed now. We haven't finished yet. We... Δεν έχουμε ολοκληρώσει, πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να πάμε στο σημείο 6. It's the working time, mm. working time mm. in the It's your report. We'll vote on the... Ψηφίζουμε λοιπόν το χρόνο εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοείας. Ονομαστική ψηφοφορία είναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για το χρόνο εργασία στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοείας. Πέρας. 39 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πριν ψηφίσουμε όμως υπάρχει μια προφορική τροπολογία από την Μαρία Ρένα. Παρακαλώ. Για λογαριασμό της κυρίας Μαρία Ρένα παρακαλώ στην υπαριθμόν 9 να διαγραφεί να διαγραφούν μάλλον οι λέξεις που είναι εντός παρενθέσεων. Εκεί που λέει δηλαδή For example, We think it's not... μέχρι και που λέει in Germany. Νομίζουμε ότι δεν είναι καλό να βάλουμε τις χώρες να βαλώνουν μεταξύ τους. Γι' αυτό προτιμούμε να διαγραφούν οι λέξεις που περιλαμβάνονται μέσα σε παρενθέσεις στο τέλος της παραγράφου. Okay, we'll... Μάλιστα. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική αυτή τροπολογία ονομαστικά. Πρόκειται περί διαγραφής. Πρόταση της κυρίας Μαρία, της Μαρία Ρένα. Mm. It's, it's a vote on, on uh, uh, the whole. Η πρόεδρος λέει ψηφίζουμε το σύνολο της παραγράφου με την τροπολογία που είναι για διαγραφή, λέει η πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε της ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Πάμε στην επόμενη αίτηση από το Βέλγιο, πάλι για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Ναι, μάλιστα. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έχουμε και τα μεταλλικά προϊόντα, κομμουνιδά Βαλενθιάνα, Κοινότητα της Βαλένθια. Ε, ψηφίζουμε την επιστολή, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, δεν ψηφίσαμε πάλι κάτι από το Βέλγιο, Κάρσιντ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεν ήταν τελευταία αυτή. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρίαση 16 Οκτωβρίου. Θα σας δω τότε. Σας ευχαριστώ για σήμερα.